Κύριε Πρόεδρε, δράτων σε ευκαιρίες για την ημερήσια διάταξη να ζητήσω επίσημα η Λέδη Άστον να έρθει στην Ολομέλεια, να έρθει στο Κοινοβούλιο να μας μιλήσει για το τι έκανε και τι θα κάνει σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στους χριστιανούς στον κόσμο. Θα θέλαμε να έρθει εδώ με μία έκθεσή της ούτω ώστε να ενημερώσει το Κοινοβούλιο λεπτομερώς επ' αυτών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, θα διεξαχθεί επίσημη συζήτηση επί του θέματος ε, την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι, λέει ο Πρόεδρος. Διαδικαστικό. Έχει το λόγο. Επικαλούμε το άρθρο 173 περί εφαρμογής του κανονισμού για να πω ότι παραβιάζεται το άρθρο 116 διότι είναι η τρίτη συνεδρίαση συνεχή συνεδρίαση τη ολομέλειας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνεται το θέμα ερωτήσει προ το συμβούλιο όπω προβλέπει το άρθρο. 116. Σα παρακαλώ δώστε μου μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό, είναι η τρίτη συνεδρίαση, πού οφείλεται και σε κάθε περίπτωση σα παρακαλώ να υπερασπιστείτε το δικαίωμα του Ευρωκοινοβουλίου και των βουλευτών να κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο και στο Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, πράγματι θα πάρουμε μια απόφαση επί του θέματος. Αυτά αφορούν τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις νέες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διότι τώρα έχουμε κοινοβούλιο δύο επιπέδων αν θέλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την άλλη. Οπότε έχουν αλλάξει οι σχέσεις. Προτείνω όμως να μην παρατείνουμε τώρα, μην ξεκινήσω τη συζήτηση τώρα, διότι όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν στο εγγύς μέλλον. Διαδικαστικό έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Δεν ξέρω εάν με παραπομπή σε μελλοντικέ αλλαγές μπορούμε να διαγράφουμε ένα κοινοβουλευτικό δικαίωμα. Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ώρα των ερωτήσεων, οπότε θα πρέπει να συνεχίζουμε μέχρι να ληφθεί μια απόφαση και όχι σε ένδειξη υπακοής να εκτελούμε κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Είναι λάθος γιατί σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άλλα ζητήματα δεν είναι ένα ανώτερο μέρος του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο πρέπει να το ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλιά σας, για αυτά που μας είπατε. Σας διαβεβαιώ ότι στην επόμενη διάσκεψη των Προέδρων, όπου εγκρίνονται οι μερίσες διατάξεις, την επόμενη πέμπτη δηλαδή, θα το θέσω το ζήτημα αυτό. Και θα δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το προσεγγίσουμε στο μέλλον. Η διάσκεψη των Προέδρων είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της ημερήσιας διατάξεως και την επόμενη πέμπτη θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ας προχωρήσουμε και ας πάμε στην ημερήσια διάταξη. Όπως λέγαμε Δευτέρα, η ομάδα των Πρασίνων, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ζήτησε τη συζήτηση με θέμα την κατάσταση στην Τινησία και να καταλήξει συζήτηση σε ένα ψήφισμα. Αυτό δεν το είχαμε σχεδιάσει προηγουμένως, δεν το είχαμε προγραμματίσει και τώρα υπάρχει πρόταση για ψήφισμα. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Μπεντίτ θέλει να το υποστηρίξει. Πιστεύω ότι το ξέρετε ότι τα γεγονότα στην νησία προχώρησαν. Δεν μπορούμε παρά να χαρούμε. Ο κύριος Μπεναλή έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Οπότε η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ τεταμένη στην Τινησία και θεωρώ ότι το κοινοβούλιο, αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει σε ένα ψήφισμα σύντομο να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι ίσω θα έπρεπε σε 6-8 εβδομάδε να διεξαχθούν εκλογέ. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε για το Φεβρουάριο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει τώρα να τοποθετηθούμε. Και γι' αυτό βάσει τη δράση μα θα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα το οποίο θα ψηφίσουμε την Πέμπτη το μεσημέρι. Καταλαβαίνω ότι δεδομένης της καταστάσεως με μεγάλο ενθουσιασμό αυτή η συνέλευση επιτέλους θα μπορέσει να ε, ψηφίσει ένα ψήφισμα, να περάσει ένα ψήφισμα για την Τινησία. Σας ευχαριστώ κύριε Κομπεντήτ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος επιθυμεί να μιλήσει υπέρ αυτής της προτάσεως. Ποιος είναι υπέρ αυτού του αιτήματος. Ε, ναι. Ορίστε. Η θέση 321. Δεν ξέρω το όνομά σας. Όχι. Ποιος θέλει να μιλήσει κατά του αιτήματο αυτού. Ορίστε. Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι το ψήφισμα θα αλλάξει την κατάσταση στην Ισία και γι' αυτό είμαι κατά. E, Οπότε θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του αιτήματο. Με ανάταση χειρός παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Απορρίπτεται το αίτημα. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Βλέπετε και η διεισόμαση ότι το αίτημα αυτό απορρίφθηκε. Επόμενη αλλαγή αφορά την πέμπτη. και συγκεκριμένα τις συζητήσεις βάσει του κανόνα 122. Η ομάδα της ε, Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Βόρειας Παράσινης Αριστεράς, ζήτησε να αποσυρθεί από την ημερήσια διάταξη η συζήτηση για τη Βραζιλία και συγκεκριμένα την έκθεση του Τσεζάρη Μπατίστη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τάβαρε, ο οποίος θα μα ε, δικαιολογήσει το αίτημα αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι συνάδελφοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να καταθέσουν ένα ψήφισμα κατά τη απόφαση της Βραζιλίας για την έκδοση του Τσέζαρε Μπατίστη στην Ιταλία, αλλά δεν είναι μια υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι το κατεπήγον, δεν είναι καν παραβίαση του κράτου δικαίου. Επιπλέον έρχεται σε μια τρομερή στιγμή όταν η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη χειρότερη, εθνική, τη χειρότερη καταστροφή στην ιστορία τη. Ο Τσέζαρε Μπατίστη είναι στη φυλακή, αναμένει την απόφαση του Ανατάτου Δικαστηρίου τη Βραζιλία, το οποίο όπως ξέρετε ε, έχει διακόψει της του. Ε, εκφράζω λοιπόν την αλληλεγγύη μου με, τα... την οικογένεια των θυμάτων και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν είμαι υπέρ της πολιτικής βίας αριστερής ή δεξιάς. Αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε την περίπτωση του Νοτίου Σουδάν ή του Σουνταρτοπίπ στην Ινδονησία ή την περίπτωση της ε, Παλαιστίνης. Θα αλλάξουμε λοιπόν την ε, τακτική μας και δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το οποίο κάνουμε συνήθω. Εγώ προτείνω να φύγει η Βραζιλία από την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο που ήθελε να εκφραστεί υπέρ του αιτήματο. Δεν βλέπω κάποιον. Θέλει κάποιος να μιλήσει κατά του αιτήματο αυτού. Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα ονόματι της ομάδας μου και πιστεύω ονόματι όλου του Κοινοβουλίου να υπογραμμίσω στεναρά το πόσο κοντά είμαστε στο λαό της Βραζιλίας για το πένθος του που σχετίζεται με τις πρόσφατες πλημμύρες. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εδώ θέλουμε να σταθούμε δίπλα τους. Και επαναλαμβάνω ταυτόχρονα ενώματι των προτινόντων και ελπίζω εκ μέρους όλου του Κοινοβουλίου την πρόθεσή μας τη στεναρή να συζητήσουμε το θέμα αυτό διότι δεν έχει αποδοθεί ακόμα δικαιοσύνη διότι η υπόθεση του Τσέζαρη Μπατίστη θα πρέπει να δικαστεί, να εξεταστεί περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να κάνει τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο να εισακουστεί στο διεθνές προσκήνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να εκφραστεί πέρα του, να τοποθετηθεί πέρα του αιτήματο αυτού. Το 652. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω το αίτημα Ταβάρες γιατί δεν είναι κάτι το κατεπήγον. Ο κύριος Μπατίστη είναι στη φυλακή. Δεν μπορούμε ε, να υποθέσουμε πως θα εξαφανιστεί. Άρα και δεν νομίζω πως θα πρέπει να ανακατευόμαστε σε υποθέσεις μεμονωμένες οι οποίες ακόμη κρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε τώρα. Ποιοι είναι υπέρ του αιτήματο το οποίο υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Ενωμένη Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, σε σχέση με την ε, συζήτηση που αφορά την έκδοση του Τσέζαρ Μπατίστη και την διαγραφή της από την διάταξη. Υπέρ, κατά, Α, ευχαριστώ πολύ, αποχές. Απορρίπτεται και αυτό το αίτημα. Λάβαμε λοιπόν τις αποφάσεις μας ό,τι αφορά την μερίσια διάταξη, οπότε ερχόμαστε στο σημείο 1 της μερίσιας διάταξης, που είναι η δήλωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Τινησία. Θα επακολουθήσει ευθύ αμέσω δήλωση της Επιτροπής και θα μιλήσουν ε, και οι πρόσωποι των πολιτικών ομάδων.